ήταν σε μια κατάσταση ιδιαίτερη θα έλεγα στην περιφέρεια αυτής. Ξέρετε ότι έχουμε σύνορα με την Βενεζουέλα. Έχουμε μια περίπλοκη ε, γειτονία με τον Ισημερινό Ήμασταν στην ε, λίστα των παραβιαστών σε εισαγωγικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του καταλόγου του, της ε, Νοτιοαμερικανικής Ένωσης όπως είπαμε και των Ηνωμένων Εθνών. Και φυσικά είχαμε και θέματα και με τις ε, χώρες της Κεντρικής Αμερικής και τα νήσους της Καραϊβικής και γι' αυτό υπήρχαν και αντιστάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την επικύρωση της συμφωνίας με την Κολοβία και το ίδιο μάλιστα είχε συμβεί και στα πλαίσια του Αμερικανικού Κογκρέσου. Εμείς προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την κατάσταση, την εξωτερική εικόνα και την εσωτερική όμως της χώρας μου. Εμείς προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε την οικονομία μας, να την ενισχύσουμε μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές και ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε 50 χρόνια ένα σύραξης, 50 χρόνια πολέμου. Ξεκινήσαμε λοιπόν μια διαδικασία διαπραγματευτική, σοβαρή, ρεαλιστική και αξιοπρεπή με ε, με τους μαχητές της ΦΑΡΚ. Στον οικονομικό τομέα μπορέσαμε μέσω νόμων που πέρασαν από το Κογκρέσο να διασφαλίσουμε την απαιτούμενη κυβερνησιμότητα της χώρας χρησιμοποιώντας το πρότυπο που είχε χρησιμοποιήσει και ο πρόεδρος Λίνκολν ο οποίος είχε προσκαλέσει ε, και τους αντιπάλους τους στις εκλογές να πάρουν μέρος της ε, στην κυβέρνηση. Έτσι διασφαλίσαμε λοιπόν ε, μια σωστή λειτουργία του Κογκρέσου της χώρας και περάσαμε νόμους, νομικούς, νόμους συγγνώμη, στον τομέα που ενίσχυσαν την οικονομία μας. Οδηγηθήκαμε σε πολύ θετικά λοιπόν αποτελέσματα με τέτοιο τρόπο που μπορούμε πλέον τώρα να πούμε ότι η Κολομβία είναι η χώρα της Λατινικής Αμερικής η οποία αναπτύσσεται με βαθμό υψηλότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της περιοχής. Είναι η χώρα η οποία έχει χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού από τις υπόλοιπες της περιοχής. Η Κολομβία είναι η χώρα η οποία έχει το μεγαλύτερο ποσοστό δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Είμαστε, ε, ε, κατεβάζουμε την ανεργία εδώ και 50 μήνες, από τον ένα μήνα στον άλλο συνεχώς. también en la parte social. Νομίζω ότι αυτό επηρέασε και τα θέματα στην κοινωνία των πολιτών. La pobreza. Προσπαθήσαμε να μειώσουμε την φτώχεια στην Κολομβία ε, και το καταφέραμε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες. Ένα τεράστιο ρεκόρ αυτό για χώρα της Λατινικής Αμερικής. Μέσα σε τέσσερα χρόνια μειώσαμε την φτώχεια σε αυτό το ποσοστό που είπα και το ίδιο επίσης και με τη λεγόμενη ακραία φτώχεια. Μία από τις βασικές μας προτάσεις ήταν να εκριζώσουμε ε, την ακραία φτώχεια από το κολομβιανό έδαφος. Και για πρώτη φορά προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τα πράγματα ε, σε περιπτώσεις ε, για τις οποίες ντρεπόμασταν. Ήμασταν οι πρωταθλητές της ανισότητας στην περιοχή αυτή, από όλες τις χώρες της περιοχής. Και προσπαθήσαμε εμείς να μειώνουμε τις ανισότητες και τώρα βρισκόμαστε στον μέσον όρο περίπου, αν και μας λείπει πάρα πολύ δρόμος ακόμα. Ε, υπάρχει πάντα πολύ μεγάλη φτώχεια στην Κολομβία, το 30% των Κολομβιανών πολιτών υποφέρουν από αυτή Έχουμε λοιπόν ακραίες μορφές ένδυας, άνω του 8% του πληθυσμού και η, απόσταση ανάμεσα στους φτωχούς και στους πλούσιους ανάλογα με την περιοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε λοιπόν πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Το πιο σημαντικό όμως είναι να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να απελευθερώσουμε το πραγματικό δυναμικό της χώρας μας και να εξασφαλίσουμε την ειρήνη στην Κολομβία μετά από 50 χρόνια συγκρούσεων, μετά από 50 χρόνια πολέμου. Ενός πολέμου που κόστισε πολύ αίμα στην Κολομβία, πολύ, οδήγησε σε μεγάλο πόνο και βάσανα. Πάνω από 6 εκατομμύρια θυμάτων κόστισε στην Κολομβία. Προσπαθούμε με ένα νόμο τον οποίο εγκρίναμε να επανορθώσουμε και να επουλώσουμε τις πληγές που δημιούργησε αυτός ο, ο πόλεμος σε, σε τόσο πολλά μέρη της Κολομβίας. Από τη στιγμή της έγκρισης αυτού του νόμου μέχρι τώρα δόθηκε επανόρθωση σε πάνω από 400.000 θύματα. Βέβαια είναι 6 εκατομμύρια τα θύματα και οι εκτοπισμένοι του πολέμου αυτού. Το πιο σημαντικό όμως είναι το να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε την ειρήνη και γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία που ξέραμε ότι θα προσκρούσει σε εμπόδια, σε δυσκολίες. Και κατανόησα κι εγώ ίδιος ότι το να επιτύχει κανείς την ειρήνη είναι πολύ πιο δύσκολο από το να διεξαγάγει τον πόλεμο και εγώ αναγκάστηκα να διεξάγω, να διεξαγάγω τον πόλεμο και με μεγάλη αποτελεσματικότητα, αλλά τώρα είναι ο καιρός της ειρήνης. Νομίζω ότι οι περιστάσεις τώρα στην Κολομβία είναι τέτοιες που ήταν έφορο το έδαφος για να ξεκινήσει μια επιτυχής διαδικασία ειρήνευσης. Εδώ και τρία χρόνια λοιπόν, τρία μισή χρόνια, ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις σε μια μυστική φάση καταρχήν με τις ε, ΦΑΡΚ, με τους ε, αντάρτες αυτούς, τις ένοπλες αυτές δυνάμεις, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή ατζέντα. Μια ατζέντα επί τη βάση της οποίας θα μπορούσαμε να έχουμε, εάν μπορούσαμε να έχουμε συμφωνία για αυτή την ατζέντα, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στη διακήρυξη του τέλους της σύγκρουσης. Αυτή η πρώτη φάση που ήταν μια φάση μυστικών διαπραγματεύσεων, απεδείχθη επιτυχής. Καταφέραμε να συμφωνήσουμε για ένα θεματολόγιο που περιλαμβάνει πέντε σημεία και μπόρεσαμε έτσι πριν από δύο χρόνια να δηλώσουμε στο Όσλο ενώπιον όλου του κόσμου ότι θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις επί τη βάση αυτών των πέντε σημείων. Έχουμε ήδη συμφωνήσει για τρία από αυτά τα πέντε σημεία. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο σημείο αφορούσε την αγροτική ανάπτυξη στην Κολομβία. Συμφωνήσαμε για μια σειρά από μέτρα τα οποία θα δώσουν τη δυνατότητα στους αγρότες της Κολομβίας και στην ύπεθρο της Κολομβίας να έχει μια ανάπτυξη, να δοθεί η απαραίτητη μέρημνα για την αγροτική ανάπτυξη στην Κολομβία. Γιατί εκεί έχει συγκεντρωθεί η στέρηση, η φτώχεια και επομένως και οι συγκρούσεις καταφέραμε να συμφωνήσουμε και σε ένα δεύτερο σημείο που είναι η πολιτική συμμετοχή. Σε βασικές γραμμές αυτό το οποίο εξασφαλίσαμε είναι μια ενίσχυση και μια εμβάθυνση της δημοκρατίας μας. Το να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα εκπροσώπησης σε περιοχές της χώρας μας που είχαν βρεθεί σε κατάσταση σύγκρουσης και οι οποίες δεν είχαν την απαραίτητη εκπροσώπηση στο, στη Βούλη της χώρας μας, το να δώσουμε περισσότερες εγγυήσεις στην πολιτική αντιπολίτευση στη χώρα μας, τελικά να κάνουμε όλα αυτά τα οποία ήταν απαραίτητα ώστε να λειτουργήσει καλύτερα η δημοκρατία στην Κολομβία. Κάτι το οποίο πρέπει να είναι μια μόνιμη άσκηση για οποιαδήποτε δημοκρατία. Συμφωνήσαμε και σε ένα σημείο το οποίο είναι μεγάλη σημασία. Ένα σημείο για το οποίο εγώ ο ίδιος επέμεινα πάρα πολύ από την αρχή να μπορέσει να συμπεριληφθεί στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων και έχει να κάνει με το εμπόριο, το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Συμφωνήσαμε με τις ΦΑΡΚ, με τους αντάρτες των ΦΑΡΚ, να εργαστούμε από κοινού. Από τη στιγμή που θα σταματούσε η ενοπλή σύγκρουση, ώστε να αντικαταστήσουμε τις παράνομες καλλιέργειες με νόμιμες καλλιέργειες. Και εργαστήκαμε από κοινού με τις ΦΑΡΚ για να μπορέσουμε να εκριζώσουμε τη λαθρεμπορία ναρκωτικών από το έδαφος της Κολομβίας. Αυτό έχει τεράστια σημασία, τεράστιες επιπτώσεις, όχι μόνο για την Κολομβία, η οποία έχει πληγεί για πάνω από 30-35 χρόνια από τη μάστιγα του λαθρεμπορίου ναρκωτικών που ήταν και το καύσιμο που κράτησε ζωντανή τη βία όλα αυτά τα 30-35 χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό πέραν της Κολομβίας για όλη την περιοχή μας, γιατί η επιτυχία που πετύχαμε να έχουμε, η σχετική αυτή επιτυχία στο να περιστύλουμε το εμπόριο ναρκωτικών στην ε, Κολομβία, το να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα καρτέλ των εμπόρων ναρκωτικού, αυτό έγινε και χάρη στην προσπάθεια των γειτόνων μας, αλλά θα είναι και προς όφελος των γειτόνων μας. Γιατί δεν έπρεπε να συμβεί αυτό που μειώνεται κατά κάποιο τρόπο σε ένα σημείο το εμπόριο ναρκωτικών και αναδύεται σε άλλα σημεία όπως γίνεται με τα συγκοινωνούντα δοχεία είχε θετικό αποτέλεσμα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου καταναλώνεται η κοκαίνη που εμείς παράγαμε. Δυστυχώς εξακολουθούμε να είμαστε ο πρώτος παραγωγός κοκαίνης στον κόσμο. Οι αντάρτες της ε, ΦΑΡΚ εξακολουθούν να προστατεύουν τις καλλιέργειες κοκαίνης, γιατί βάζουν νάρκες γύρω από αυτές τις καλλιέργειες ώστε όταν η αστυνομία ή ο στρατός πηγαίνει και προσπαθεί να εκριζώσει αυτές τις καλλιέργειες έχουν να αντιμετωπίσουν τις νάρκες. Και υπήρξαν χιλιάδες θυμάτων λόγω αυτής της ε, πρακτικής που ακολούθησαν οι ΦΑΡΚ και πολλά άτομα τα οποία έχασαν όχι είτε τη ζωή τους ή ακροτηριάστηκαν. Και επίσης υπήρξαν πάρα πολλοί οι οποίοι απλώς σκότωναν τους ε, στρατιώτες ή τους αστυνομικούς που πηγαίναν να εκριζώσουν τις καλλιέργειες κόκας. Τώρα όμως οι ΦΑΡΚ έχουν συμφωνήσει με την κυβέρνηση να υπάρξει η εκρίζωση αυτών των καλλιεργειών και να, γίνουν, να μετατραπούν αυτές οι καλλιέργειες σε καλλιέργειες οι οποίες έχουν νόμιμο χαρακτήρα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη σημαντική συμφωνία. Μένουν δύο σημεία τα οποία είναι πολύ δύσκολα παραμένει το θέμα της μεταβατικής δικαιοσύνης. Πώς θα αντιμετωπιστούν τα θύματα. Εγώ από την αρχή ζήτησα να τεθούν τα θύματα στο κέντρο της λύσης αυτής της ε, σύγκρουσης. Αυτό δεν έχει γίνει σε καμία άλλη διαδικασία ειρήνευσης. Γιατί το έκανα αυτό, γιατί το ζήτησε αυτό. Γιατί έχουμε ένα τόσο μεγάλο αριθμό θυμάτων στην Κολομβία που αν δεν ανακτήσουν τα δικαιώματά τους αυτά τα θύματα, αν δεν τους αποδοθεί ε, δικαιοσύνη, δεν θα μπορέσει μια ειρήνη να διαρκέσει. Και το νέο αυτό σχήμα δικαιοσύνης που ονομάζεται μεταβατική δικαιοσύνη είναι αυτό το οποίο μόνο θα μπορούσε να δώσει ικανοποίηση στα θύματα που δίνει πραγματικά στα θύματα το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στην αλήθεια, στη δικαιοσύνη, στην επανόρθωση και κυρίως στην μη επανάληψη όλων αυτών των κακών που έλαβαν χώρα. Την εγγύηση ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα τηρηθούν σε οποιαδήποτε λύση που θα δοθεί σε αυτήν την σύραξη στην Κολομβία. Κάναμε λοιπόν ένα τολμηρό, ένα βήμα χωρίς προηγούμενο να ζητήσουμε και να προσκαλέσουμε τα θύματα αυτά να έρθουν ενώπιον των διαπραγματευτών στην Αβάνα. Γιατί? Γιατί αν πρόκειται να σεβαστούμε τα δικαιώματα των θυμάτων, είναι τα ίδια τα θύματα τα οποία είναι οι καλύτεροι συνομιλητές μας, είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να μας πούν πώς ακριβώς θα πρέπει να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά τους. Γιατί επίσης είμαστε και η πρώτη χώρα η οποία προσπαθεί να επιλύσει μια ένοπλη σύγκρουση μέσα από το πλαίσιο της Συμφωνίας της Ρώμης. Δημιουργούμε λοιπόν ένα προηγούμενο. Οποιαδήποτε δράση στην οποία προχωρούμε, την παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον η διεθνή κοινότητα και όλες οι άλλες χώρες που έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Το να μπορέσουμε να δώσουμε ικανοποίηση στα θύματα και να του ξαναδώσουμε τα δικαιώματά τους είναι αυτή τη στιγμή το μεδούλι της επίλυση και της υπέρβασης αυτής της σύγκρουσης. Ορισμένοι νομίζουν ότι εμείς διαπραγματευόμαστε για τα δικαιώματα των θυμάτων. Όχι, είναι αδιαπραγμάτευτα τα δικαιώματα των θυμάτων. Απλώς ακούμε την άποψη των θυμάτων για να δούμε πώς μπορούμε να επιτύχουμε την ικανοποίηση των δικαιωμάτων τους με το τέλος της σύγκρουσης. Το πέμπτο σημείο το οποίο παραμένει και πρέπει να τύχει διαπραγμάτευσης είναι το λεγόμενο DDR. Η κατάθεση των όπλων, ο αφοπλισμός και η επιστροφή όλων αυτών των κατόχων στην πολιτική ζωή. Αν υπάρξει συμφωνία στα δύο τελευταία σημεία, τότε νομίζω ότι θα τερματιστεί πλέον και ο εμφύλιος. Εμείς κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να καταφέρουμε να συνδυάσουμε τις προσδοκίες από τη μία της διεθνούς κοινότητας ε, με τις προσδοκίες του Κολομβιανού λαού και τις απαιτήσει του νομικού μας συστήματος και του συντάγματός μας με τις επιθυμίες από την άλλη της ΦΑΡΚ ε, για το θέμα της λεγόμενης μεταβατικής δικαιοσύνης. Εμείς λοιπόν γι' αυτό Θέλουμε στήριξη και ζητάμε αυτή τη στήριξη από τον κόσμο και από την Ευρώπη. Θέλουμε αυτή την πολιτική μόχλευση για να μπορέσουμε να πάρουμε τις πολιτικές αποφάσεις που θα μας οδηγήσουν στην ειρήνη. Μια ειρήνη διαρκή και ε, βιώσιμη. Με ζήτησαν τι γίνεται με μια άλλη ομάδα, πολύ μικρή, που και αυτή βρίσκεται εδώ και 50 χρόνια στον πόλεμο είναι το LLN, ο στρατός της Εθνικής Απελευθέρωσης όπως λέγεται. Μια άλλη ανταρτική ομάδα. Η απάντηση σε σχέση με το LLN είναι η εξής. Βρισκόμαστε στην πρώτη φάση, την λεγόμενη μυστική φάση. Αντίστοιχη με αυτήν την οποία βιώσαμε στην αρχή με τους ΦΑΡΚ. Και γι' αυτό στην παρούσα λοιπόν φάση δεν μπορώ εγώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες για τις επαφές τις οποίες έχουμε με το LLN. Πάντως θέλουμε εμείς να έλθει η ειρήνη και να υπογράψουμε συμφωνία και με τις δύο αυτές ανταρτικές ομάδες και να μπορέσουμε σε μια κάποια φάση να ενοποιήσουμε τις διαπραγματεύσεις με τις δύο αυτές ομάδες. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος, αλλά φυσικά κάθε φάση έρχεται στον καιρό που πρέπει. Θα ήθελα να φτάσω στο τέλος λέγοντας πολύ απλά ότι η ειρήνη στην Κολομβία, για την Κολομβία, θα είναι κάτι το τρομερό. Διότι τα αποτελέσματα, οι επιπτώσεις αυτής της σύγκρουσης, της εμφύλιας ήσαν καταστροφικές εμείς παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να πετύχουμε πολλούς δείκτες κοινωνικούς και οικονομικούς μεσούσεις αυτής της σύραξης. Φανταστείτε πώς θα ήταν η χώρα μας αν δεν υπήρχε αυτή η, ε, ε, κρίση, ο εμφύλιος. Θα ήμασταν άνω του 2% σε ετήσια βάση ανάπτυξης αν είχαμε υπογράψει την ειρήνη παραπάνω από αυτήν που σημειώνουμε τώρα. Θα είχαμε αυξήσει γενικά, θα είχαμε βελτιώσει όλους τους δείκτες κατά πάνω από το 4%. Δεν έγινε βέβαια αυτό. Παρ' όλα αυτά οι αλλαγές έχουν δημιουργήσει προβλήματα λόγω της σύραξης σε πολλά τμήματα του πληθυσμού έχουν οδηγήσει σε μετακινήσεις ε, του πληθυσμού, έχουν δημιουργήσει προβλήματα ε, στις φτωχογειτονιές γύρω από τις πόλεις, προβλήματα υγείας, παθολογικά, ψυχολογικά και γι' αυτό ακριβώς επιδιώκουμε την ειρήνη. Και για πρώτη φορά εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια κάποια επιθυμία από την άλλη πλευρά, από τους συνομιλητές μας. Το αναγνωρίζω αυτό. Επίσημα και με σοβαρό τρόπο αποδέχεται κάτι το οποίο δεν είχε αποδεχθεί ποτέ στο παρελθόν και διαπραγματεύεται νομίζω με σοβαρό τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν είμαι αισιόδοξο ότι πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία εφόσον ακολουθήσουμε την κατεύθυνση την οποία έχουμε ήδη ε, πάρει. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει χρειαζόμαστε και την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητος που είναι μία από τις προϋποθέσεις που θα πρέπει όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον να είναι παρούσα. Είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία της διεθνούς κοινότητας σε μια τόσο δύσκολη διαδικασία. Εν τέλει θα έλεγα το εξής. Το μέρισμα της ειρήνης στην Κολομβία για την Ευρώπη είναι πάρα πολύ θετικό όχι μονάχα σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα το οποίο θα προέκυπτε για την ε, μείωση της προσφοράς κοκαίνης στις πόλεις της Ευρώπης, πολλές από τις οποίες βλέπουν να ανεβαίνει η κατανάλωση, αλλά επίσης και σημαντική επίπτωση για τα θέματα του περιβάλλοντος. Η Κολομβία είναι μια από τις πιο πλούσιες χώρες σε ό,τι αφορά την βιοπικιλότητα. Είμαστε η πιο πλούσια χώρα του κόσμου σε ό,τι αφορά την βιοπικιλότητα με τετραγωνικό χιλιόμετρο. Έχουμε το τροπικό δάσος, το οποίο είναι ιδιαίτερα πλούσιο από αυτή την έποψη. Έχουμε υδάτινους πόρους όπως πολύ λίγες χώρες στον κόσμο. Όλα αυτά έχουν θυγεί πάρα πολύ αρνητικά από την σύγκρουση, από τον εμφύλιο, η παράνομη εξόριξη ε, ε, μετάλλων και άλλων ορυκτών έχει και αυτή παίξει ένα πολύ αρνητικό ρόλο τροφοδοτώντας τον, τον εμφύλιο. Θα πάρουμε λοιπόν ένα σημαντικό μέρισμα σε επίπεδο περιβάλλοντος όχι μόνο για μας την Κολομβία αλλά και για όλο τον κόσμο θα είναι πολύ πιο εύκολο να μειώσουμε την αποψήλωση που ήταν το αποτέλεσμα της ε, ζήτησης που υπήρχε για την καλλιέργεια ναρκωτικών και ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σε μια οικονομία η οποία θα έχει μηδενική καθαρή εκπομπή διοξιδίου του άνθρακος το 2020 και ελπίζουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε αυτό το στόχο ακόμα νωρίτερα. Γι' αυτό η διαδικασία αυτή της ειρήνευσης στην Κολομβία είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να δώσει τέρμα στη μοναδική ενοπλή σύγκρουση που συνεχίζεται στο, διεθνέ, στο δυτικό ημισφαίριο. Είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία και πρέπει να έχει την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας και είναι απαραίτητη η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πάρει ευτυχώς αυτή την ε, υποστήριξη. Δεν μπορώ παρά να έχω λόγια ευγνωμοσύνη σε εσά για αυτή την υποστήριξη και τώρα στην τελική φάση των διαδικασιών αυτών χρειαζόμαστε αυτή την πολιτική υποστήριξη η οποία θα μας δώσει την απαραίτητη νομιμοποίηση για να λάβουμε τις οριστικές αποφάσεις οι οποίες θα θέσουν τέρμα σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο μεταξύ των τέκνων ενός και του ίδιου έθνους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι η έκκλησή σας είναι μια έκκληση η οποία θα έχει ανταπόκριση σε εμά, θα έχετε την υποστήριξή, υποστήριξή μας. Η σε αυτή γίνεται μαζί με την αντιπροσωπεία για τις χώρες του Συμφώνου των Άνδεων, όπου προεδρεύει ο κύριος Τεγκράντες Πασκουάλ στον οποίο θα ήθελα εν συντομία του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας της Κολομβίας, θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω και τον ε, πρεσβευτή της Κολομβίας με τον οποίο έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές. Ως πρόεδρος της ε, αντιπροσωπείας για τις ε, χώρες των Άνδελ είχα την ευκαιρία να συναντηθώ πολλές φορές με εκπροσώπους της χώρας σας. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά τα οποία σίγουρα θα θίξουν αυτοί οι οποίοι θα λάβουν το, το λόγο θα αναφέρουν, όπως είναι οι πολυ, πολυμερείς συμφωνίες με την Κολομβία. Θα ήθελα να τονίσω όμως κάτι το οποίο κατά την άποψή μου είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την τωρινή κατάσταση της Κολομβίας, κατά την άποψή μας. Θα πρέπει να διεκδικήσουμε τα εύσημα κατά κάποιο τρόπο για τον ειδικό ρόλο που έπαιξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις προξενικές θεωρήσεις. Ξέρετε ότι στις 29 του προηγούμενου μηνός η Κομισιόν ενέκρινε μια έκθεση όπου υπήρχε θετική κρίση σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση όλων των προαπαιτουμένων. Με την απόφαση αυτή υπήρξε μια αναγνώριση της προόδου στα οικονομικά θέματα, του σεβασμού των θεμάτων υπηκότητα στην, στην ε, Κολομβία και λέω ότι εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο γιατί εμείς προωθήσαμε αυτήν την ταχεία διαδικασία η οποία μπόρεσε να φτάσει στο επίπεδο της ε, Κομισιόν και του Συμβουλίου που πρέπει να πάρει την τελική απόφαση. Ελπίζουμε ότι το πρώτο τρίμηνο το Συμβούλιο θα πάρει την απαραίτητη απόφαση η οποία θα μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο τρίμηνο του 2015. Επομένως με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει η δυνατότητα ε, προξενικών θεωρήσεων βραχίες διάρκειας στην χώρα του Σέγγεν, όπως έγινε προηγουμένως με το Περού. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για τη σημαίνει Κολομβία. Η οικονομική ανάπτυξη που επετέφθη έχει προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις, δημιουργεί μια νέα μέση τάξη στην Κολομβία που οδηγεί και μεγαλύτερη ασφάλεια και στη χώρα αυτή και στην περιφέρεια της Κολομβίας και επίσης και για τους επενδυτές και τον οικονομικό κόσμο. Το να περάσετε από τον κύκλο των βασάνων, του θανάτου και της βίας, το να περάσετε σε ένα κόσμο ο οποίος είναι ένας κόσμος ασφάλειας, δικαίου και ένα έφορο επιχειρηματικό κλίμα, μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ένα τρίτο στοιχείο είναι να εξασφαλιστεί η ποιότητα της δημοκρατίας και του, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να υπάρχει σε μια χώρα όπως η δική σας η ατιμορρησία. Η διαδικασία ειρήνης δεν προβλέπει την ατιμορρησία. Προβλέπει ένα διάλογο ο οποίος θα έχει πράγματι ε, αποτελέσματα θετικά. Ναι, θα είμαι σύντομος. Αυτά που είπατε είναι ότι θέλετε να αλλάξετε τα όπλα, τα όπλα που να γίνουν ψήφοι και η καλλιέργεια κόκας να γίνει καλλιέργεια νόμιμων προϊόντων. Έχετε διαλέξει το δρόμο της ειρήνης, τον δρόμο του διαλόγου. Με τον τρόπο αυτό έχετε κάνει κάτι το οποίο είναι υποδειγματικό, το οποίο πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς για τις άλλες χώρες του κόσμου. Είναι αυτή η Κολομβία και είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, της δικαιοσύνης χωρίς ατιμορρησία που χαρακτηρίζει την Κολομβία του Προέδρου Σάντος. Πιστεύουμε ότι είναι ένα υπόδειγμα για όλους και εγώ θα ήθελα να σας πω ότι είναι το μοντέλο το οποίο θα ήθελα να δω να επικρατήσει όλη την Αλληνική Αμερική. Ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε να συνεχίσουμε λοιπόν στη θέση του Προέδρου. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Λάγκε, ο οποίος είναι Πρόεδρος της ε, Αντιπροσωπείας και εισηγητής. Ja, danke Σας ευχαριστώ, λέει ο κύριος Λάγκε. Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που σας συναντώ και πάλι εδώ. Είχαμε στο παρελθόν να συναντηθούμε στην Κολομβία πολλές φορές για την εμπορική συμφωνία και ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου και προηγουμένως ως εισηγητής για την εμπορική αυτή συμφωνία Χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι μπορέσαμε να έχουμε μια συμφωνία για τις αρχές της εμπορική αυτής συμφωνία που θα οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη για την Κολομβία και η οποία ήδη έχει πραγματοποιηθεί από το 2012 μέχρι σήμερα. Και πέραν αυτής τη συμφωνίας έχουμε ένα οδικό χάρτη για τη βελτίωση της αηφορίας και της σταθερότητας των σχέσεών μας και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι μπορέσαμε να έχουμε αυτή τη συμφωνία να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένα βήματα για τη σταθεροποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης στην Κολομβία. Τελευταία ήμουνα το Μάρτιο του έτου αυτού στην Κολομβία και εγώ έχω χαιρετήσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι μπορέσαμε να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά και ότι μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά στοιχεία αυτή τη διαδικασία. Ξέρω ότι δεν βρισκόμαστε στο τέλο μια διαδικασία, αλλά στην αρχή μια διαδικασία που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού. Και εδώ πέρα περιλαμβάνεται και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Εδώ θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο και η διαδικασία ειρήνευση, γιατί όπω αναφερθήκατε υπάρχουν οι μελέτε αυτέ που δείχνουν το μέρισμα τη ειρήνη θα μπορέσει με την η ειρήνη αυτή να έχει μεγαλύτερη ζωτικότητα η εμπορική συμφωνία με την Ευρώπη και να δημιουργήσει περισσότερη οικονομική ανάπτυξη για την χώρα σας, αλλά συγχρόνως αυτή η εμπορική συμφωνία μπορεί να παίξει ένα θετικό ρόλο για την σταθεροποίηση της διαδικασία ειρήνης, γιατί θα αναπτύξει καλύτερες οικονομικές ε, δυνατότητες στη χώρα αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε το διάλογο και τη συνεργασία και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η διαδικασία ειρήνης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό δομικό λίθο για το μέλλον της χώρας σας. Έχω εδώ μια έκθεση του Ιδρύματος Φρίντριχ Έμπερτ, η οποία είναι πολλές φορές, υπήρξε πολλές φορές επικριτική σε σχέση με τη χώρα σας, αλλά εδώ ο τίτλος είναι «Η Κολομβία αποφασίζει να ακολουθήσει το δρόμο της ειρήνης». Αυτό είναι ένα πραγματικά σημαντικό μήνυμα το οποίο είναι σημαντικό για όλους μας για να υποστηρίξουμε σε μια ευρεία συμμαχία αυτήν τη διαδικασία ειρήνευσης ώστε να μην υπάρξουν οι και μέσα στα πλαίσια αυτά είναι πάρα πολύ σημαντική η εμπορική συμφωνία. Ευχαριστώ. Έχουμε 15 ομιλητές, σας παρακαλώ να είσαστε σύντομοι για να έχουμε τη δυνατότητα να τελειώσουμε εγκαίρως και με πήρε τηλέφωνο προηγουμένως η κυρία Μογκερίνη και με πληροφόρησε ότι για την περίπτωση του, ε, του Κωσόβου θα λάβει χώρα μια ανεξάρτητη έρευνα. Ο κύριος Μίλαν Μόν έχει το λόγο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του οποίου είμαι συντονιστής, να σας καλωσορίσω, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας της Κολομβίας. Είναι μεγάλη τιμή για μας και η παρουσία σας εδώ είναι θα έλεγα και σύμβολο της εξαιρετικής σχέσης την οποία έχει η χώρα σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η παρουσία σας εδώ αναγνωρίζει τον ρόλο, τον πρωτοποριακό τον οποίο εμείς παίξαμε για την εντατικοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ε, στην Δημοκρατία της Κολομβίας. Ε, παίξαμε ρόλο και ε, για την επικύρωση φυσική της τελικής συμφωνίας ανάμεσα στα δύο μέρη και νομίζω ότι αυτή η συμφωνία βοήθησε πάρα πολύ στην ανάκαμψη της οικονομίας. Η διμερής συνεργασία επίσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κολομβία και η λεγόμενη ρήτρα phasing out σε οικονομικό επίπεδο βοηθά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον και τη χώρα σας. Και όπως είπε και ο Πασκουάλ Ντε Γράντες, βοηθήσαμε έτσι ώστε να υπάρξει η εξέλιξη αυτή θετική η οποία στο μέλλον άμεσα θα έλεγα και ελπίζω να δώσει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα η οικονομία σας είναι μία από τις ισχυρότερες της περιοχής, η απασχόληση από τις υψηλότερες, ο πληθωρισμός από τους χαμηλότερους ή αν όχι ο χαμηλότερος στην Λατινική Αμερική και φυσικά υπάρχει το θέμα της ακραίας φτώχειας την οποία προσπαθείτε να καταπολεμήσετε και εσείς ε, τα ποσοστά που μας δώσατε είναι πράγματι εντυπωσιακά. Έχετε μια μεταρρυθμιστική τάση και δράση Ελπίζω να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση στην τρομακτική προσπάθεια την οποία κάνετε και θα ήθελα να μας πείτε κύριε Πρόεδρε τι περιμένετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι περιμένετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Επιτροπή μας την Κοινοβουλευτική των Εξωτερικών Υποθέσεων. Είναι μια πολύ επίσης ε, ε, σημαντική χώρα και στα πλαίσια της λεγόμενης Συμμαχίας του Ειρηνικού τι μπορείτε να μας πείτε για την παρούσα κατάσταση της συνεργασίας αυτής. Είμαι βέβαιος ότι ο επόμενος συνάδελφος θα, θα είναι πιο γρήγορος και από σας. Χαιρετίζω την παρουσία σας κύριε Πρόεδρε και ελπίζω η σημερινή μας συνάντηση να δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να παίξει έναν πιο ενεργό ρόλο για την ε, ειρηνευτική διαδικασία στη χώρα σας που ελπίζουμε να πετύχει. Και σε αυτό το πνεύμα, γνωρίζοντας ότι είναι πολλοί φραγμοί, υπήρξαν πολλοί φραγμοί για την ειρήνευση της χώρας, θα ήθελα να αναφέρω τη δυνατότητα πολλών πολιτικών που αναφέρουν στη χώρα μας την ιδέα μιας και χειρίας στην Κολομβία έχει γίνει αυτή η πρόταση και τι έχετε να μας πείτε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς αυτήν τη δυνατότητα που θα μπορούσε να είναι μια πρώτη γεύση της μελλοντικής ειρήνης. αυτά που μας είπατε για τα δικαιώματα των θυμάτων το με βρίσκουν σύμφωνο, αλλά λίγο μόλις μέρες πριν η αντιπροσωπεία των θυμάτων στις συζητήσεις της Αβάνας φαίνεται ότι έλαβαν απειλές, θανατικές απειλές. Τι έχετε λοιπόν να πείτε ως τη δυνατότητά σας <laughs> να διασφαλίσετε ότι τα θύματα και οι εκπρόσωποι τους δεν θα παρουσιαστούν απλώς στην Αβάνα αλλά θα παίξουν σημαντικό ρόλο πραγματικά στις συζητήσεις και ότι δεν θα ακουστούν μόνο λόγια για τις αποζημιώσεις τους στην Αβάνα αλλά θα υπάρξουν και έργα. Τι προστασία θα τους χορηγήσετε αφού έχουν ήδη υπάρξει θανατικές απειλές. Τώρα για την ασφάλεια. Η υπάτη Αρμοστία για τα ανθρώπινα δικαιώματα λέει ότι δυστυχώς η Κολομβία ήταν, στην Κολομβία η τελευταία δεκαετία ήταν χειρότερη για, ως προς τις δολοφονίες των αγωνιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ΙΕ λέει ότι είναι πάνω από 95% ο δείκτης τέτοιων εγκλημάτων. Με όλα αυτά στο μυαλό μας, ο προϋπολογισμός για την προστασία ανθρώπων, για σωματοφύλακες και για συνδικαλιστές έχει περικοπεί κατά θα επανέλθετε στα προηγούμενα ποσά και τέλος. Μία επιτυχής ειρηνευτική διαδικασία όχι μόνο αποζημιώσεις για τα θύματα αλλά πραγματική την αποκατάσταση για τις ε, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τι έχει γίνει. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Τώρα οι συντονιστές για δύο λεπτά και μετά οι υπόλοιποι για ένα λεπτό. Ο δόκτωρ Τάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματο συντηρητικών σα συγχαίρω για την επανεκλογή σα τον Ιούλιο ω Πρόεδρο τη Κολομβία για δεύτερη φορά. Ακόμη θυμάμαι τη... όταν πήγα στον ε, παλάτι Ναρένιο και είχα τότε αναλάβει μια καμπάνια για την εμπορική συμφωνία του Περού, της Κολομβίας και της Ένωσης εγώ είμαι γνωστός φίλος της Κολομβίας και θαυμάζω ιδιαίτερα και τον προκάτοχό σας, τον πρόεδρο Ουρίβε, στην προσπάθειά του να νικήσει κατά τον ΦΑΡΚ στρατιωτικός. Επίσης, ίσως πετύχατε ένα μικρό οικονομικό θαύμα που πολλοί δεν πίστευαν ότι μπορεί να υπάρξει καν. Με μεγάλη χαρά άκουσα ότι η ανάπτυξη θα είναι γύρω στο 5% πάνω και από το γειτονικό Περού. Και αυτό είναι άξιο συγχαρητηρίων. Και επίσης χαίρομαι για την πιθανή λήξη των δεκαετιών ε, σύραξης με τις ΦΑΡΚ, με τους αντάρτες. Ελπίζω πραγματικά η ειρήνη αυτή, η ειρήνευση αυτή να φέρει και τα οικονομικά της αποτελέσματα. Δύο ερωτήματα θέλω να θέσω. Το ένα, ελπίζοντας την ειρήνευση με τη ΦΑΡΚ, τι θα γίνει με τον γείτονά σας στη Βενεζουέλα. Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος Μαδούρο μπορεί να είναι χειρότερος και από τον Τσάβες και οι σχέσεις σας δεν ήταν πάντοτε ήσυχες. Δεύτερον, για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Στη χώρα μου γίνεται συζήτηση και σε άλλες χώρες της Ένωσης για το κατά πόσον η απελευθέρωση των ναρκωτικών, όχι μόνο των μαλακών όπως της Κανάβεως, αλλά και των άλλων, δεν προτείνεται. Τι φρονείτε εσείς για μια απελευθέρωση των ναρκωτικών για κατάργηση της απαγόρευσής τους δηλαδή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή, Πρόεδρε Σάντος, να σας ξαναβλέπω. Πριν από ένα χρόνο, μια ομάδα φιλελευθέρων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από αλλού σας επισκέφθη και μας εντυπωσίασαν πολλά πράγματα. Οι πολιτικές σας για το περιβάλλον, οι κοινωνικές πολιτικές και οι οικογενειακός προγραμματισμός και φυσικά και η διαπραγματεύση για την ειρήνευση. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς αυτές οι ειρηνευτικές συνομιλίες μπορούν να οδηγήσουν σε μια διαρθρωτική ειρήνη. Είπατε εσείς είστε δεσμευμένοι και η ΦΑΡΚ επίσης, αλλά υπάρχουν και άλλες οργανώσεις ένοπλες. Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε μαζί με τη ΦΑΡΚ μια ειρήνη όλου του έθνους Κολομβίας με τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να σας ε, ευχαριστήσω Πρόεδρε Σάντος που ήρθατε και μας δώσατε την ευκαιρία να ακούσουμε τα λόγια σας που μας δίνουν μεγάλη ελπίδα και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη διαδικασία αυτή της Σαββάνας. Είμαι ειλικρινής όμως, έχουμε πολλές ανησυχίες γιατί και η ιστορία της χώρας σας μας δίνει πάρα, πολύ, ε, πάρα πολλούς λόγους ε, ανησυχίας. Μια πατριωτική ενέργεια από πολλούς θεωρήθηκε ότι ήταν μια γενοκτονία και υπήρξαν πάρα πολλές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εφέτος έχουμε το, ακόμα στην Κολομβία το ρεκόρ για φόνους συνδικαλιστών. Λέτε ότι βελτιώνεται το σχήμα προστασίας όλων αυτών, αλλά δεν έχουμε δει ακόμα τα αποτελέσματα. Επίσης το θέμα της δικαιοσύνης ε, που ακόμα δεν έχει ικανοποιητικό χαρακτήρα. Υπάρχουν όχι μόνο τα θύματα, αλλά υπάρχει και το θέμα της ιδιοκτησίας των γεών και τα θέματα των παραστρατιωτικών οργανώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σας υποστηρίξει, αλλά πρέπει να σας υποστηρίξει με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τον τρόπο αυτό επίσης ότι θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν οι δομικές ρίζες αυτής της σύγκρουσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν θα δοθεί ικανοποίηση στα θύματα και θα επανέλθουν οι αυτόχθονες κοινότητες στις γέες τους. Ερωτήματα για να κλείσω. Ποια ε, μέτρα θα πάρετε ε, έναντι των, ε, της συστηματικής παρακολούθησης από τις μυστικές υπηρεσίες της Κολομβίας έναντι των δημοσιογράφων, ακόμα και των μελών της κυβέρνησης που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις. Δεύτερον, μήπως πιστεύετε ότι δεν έχει νόημα να έχετε διαπραγματεύσεις με τις ε, ΦΑΡΚ και διερευνητικές ε, συνομιλίες με την ΕΛΕΝΕ που είναι οργανώσεις που η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι είναι τρομοκρατικές οργανώσεις και η οικολογία επίσης. Μήπως θα πρέπει να αλλάξει αυτό για να μπορέσει να επικρατήσει η ειρήνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο ήδη αναφέρθηκε. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών. Κάτι το οποίο θα σας απασχολήσει στα πλαίσια της επίσκεψής σας στις Βρυξέλλες. Εμείς ε, θεωρούμε ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία. Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη βέβαια ε, συνθήκη δεν έχει βελτιώσει την κατάσταση των παραγωγών καφέ σαν παράδειγμα. Ένα παράδειγμα του πληθυσμού που δεν έχει επηρεαστεί θετικά. Και δεν έχει μειωθεί το παράνομο χρήμα το οποίο κυκλοφορεί λόγω του παράνομου εμπορίου ε, ναρκωτικών, λαθρεμπορίου ναρκωτικών κτλ. Και τα πράγματα χειροτερεύουν γιατί ακόμα και όταν παρεμβαίνουν μεγάλες επιχειρήσεις βασική τους μέρημνα είναι να αποφύγουν την πληρωμή φόρων. Και γι' αυτό θα ήθελα να μας αξιολογήσετε τα αποτελέσματα της συμφωνίας που υπογράψατε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μας πείτε αν έχετε ξεκινήσει διάλογο για να δείτε τι είναι τα πράγματα τα οποία θα πληθείτε να βελτιώσετε στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ξεκινώντας να απαντήσω στον κύριο Βιγιάν για το τι ελπίζει η Κολομβία, τι περιμένει μάλλον η Κολομβία από την Ευρώπη. Και επίσης να σας μιλήσω και για την λεγόμενη συμφωνία του ειρηνικού, η συνεργασία του ειρηνικού. Εμείς αυτό το οποίο συζητάμε εδώ με την επίσκεψή μας στην Ευρώπη είναι η λεγόμενη πολιτική στήριξη. Εμείς καλούμεθα να πάρουμε ορισμένες αποφάσεις πάρα πολύ δύσκολες, οι οποίες είναι πάρα πολύ πιθανό ότι δεν θα ικανοποιήσουν όλους και δεν θα ικανοποιήσουν απόλυτα κανένα. Οι διαπραγματεύσεις αυτές πάντα στο τέλος αφήνουν όλο τον κόσμο ε, λίγο ανικανοποίητο αλλά προσπαθούμε να συνδυάσουμε και τις προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα προηγούμενο θα έλεγα επιζητώντας την εφαρμογή των νόμου και της δικαιοσύνης κάτι το οποίο ε, είναι, το βλέπουν διαφορετικά αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη να μην λειτουργήσει σαν εμπόδιο για την ειρήνη. Αλλά νομίζω ότι εμείς επιδιώκουμε την ειρήνη και γι' αυτό ακριβώς συζητάμε μια ισχυρή πολιτική στήριξη από την Ευρώπη. Τώρα σε πιο συγκεκριμένο επίπεδο εμείς ε, στην ουσία διαρθρώνουμε στην παρούσα φάση μια μεγάλη σειρά προγραμμάτων για τις περιοχές οι οποίες έχουν καταστραφεί από την σύραξη, δηλαδή εναλλακτικές καλλιέργειες ε, ε, μετατροπής των, των ανταρτών σε δασοφύλακες. Νομίζω ότι Ξέρουμε ότι έτσι μπορεί να υπάρξει μια σωστή διαχείριση των ε, τροπικών δασών της χώρας. Ε, νομίζω ότι αυτά είναι παραδείγματα τα, στα οποία η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα για τη συνεργασία του ειρηνικού. Μπορώ να πω με πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι βρισκόμαστε σε μια στην πιο απαιτητική αν θέλετε μορφή λατινοαμερικανικής συνεργασίας χωρών της Λατινικής Αμερικής. Είχαμε μια επικοινωνία και με, στα πλαίσια μια συζήτηση με τον πρόεδρο του Περού, τον Αλαν Γκαρσία, ε, αυτή την επικοινωνία και με τους πρόεδρους του Μεξικού και της Χιλής το μετατρέπουμε σε ένα σχέδιο φιλόδοξο, πρακτικό, χωρίς πάρα πολλά γραφειοκρατικά βαρύδια, αλλά κάτι το οποίο είναι ευέλικτο και μπορεί να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις και να επιτρέψει ε, θα έλεγα τη συνεργασία ανάμεσα στις τέσσερις χώρες με τα καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα στην Λετινική Αμερική. Εμείς δεν είμαστε ανταγωνιστές με τη Βραζιλία, προσπαθούμε ε, να έχουμε όμως, έχουμε μάλλον. Ευρώπη κατά κεφαλήν εισόδημα ανώτερο από, από το αντίστοιχο της Βραζιλίας και προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις οικονομίες μας συνδυάζοντας έτσι τις δυνάμεις μας γιατί ο συνδυασμός των δυνάμεων μας θα μας κάνει ακόμα πιο ισχυρούς. Υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες είναι παρατηρητές, παρατηρήτριες αν θέλετε. Υπάρχουν 29 χώρες οι οποίες βλέπουν το τι κάνουμε και ακριβώς η διαδικασία αυτή είναι μια φιλοδοξία θα έλεγα πάρα πολύ απαιτητική. Τώρα έρχομαι σε αυτά που έλεγε ο κύριος ε, ε, Χάουιτ σχετικά με την κατάπαυση του πυρός. Θα ήθελα να πω εδώ ότι ε, αυτό είναι εγώ είμαι υπεύθυνος γι' αυτό. Εγώ έθεσα σαν προϋπόθεση της έναρξης των διαπραγματεύσεων να μην ξεκινήσουμε το θέμα της κατάπαυσης του πυρός παρά μόνο στο τέλος της διαδικασίας. Για ποιο λόγο? Πρώτον, γιατί η εμπειρία μέχρι τώρα μας έχει δείξει ότι στα πλαίσια μιας τόσο σύνθετης εδαφικής πραγματικότητας όπως αυτή της Κολομβίας, αυτό το οποίο συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις είναι να συγκεντρώνουμε ένα μεγάλο ποσοστό των συζητήσεων στα διαχειριστικά θέματα της κατάπαυσης του πυρός. Ενώ ε, και μάλιστα η άλλη ομάδα, η Ανταρτική, το LLN δεν συμμετέχει έτσι κι αλλιώς σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτή τη φάση. Τώρα από την άλλη η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι οι ΦΑΡΚ είναι πάρα πολύ ικανές να επιδιώκουν ε, της καταπαύσης του πυρός για να ενισχύονται στρατιωτικά και πολιτικά. Ε, και τρίτον, αυτή η διαδικασία λειτουργεί με στρεβλό τρόπο και ε, δίνει τη δυνατότητα στις ένοπλες δυνάμεις των ΦΑΡΚ να διαπραγματεύονται χωρίς καμία στρατιωτική πίεση. Είναι κάτι το οποίο πήρα σαν απόφαση και μου κόστισε πολιτικά το να μην προσυπογράψω την κατάπαυση του πυρός. Εγώ έχω πάει, συζητώ, διαπραγματεύομαι στην Αβάνα και με κατηγορούν ότι κάνω πόλεμο στην Κολομβία ταυτόχρονα. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο δρόμος που ακολουθώ είναι ο συντομότερος για να τερματιστεί η συγκεκριμένη σύραξη και αυτός είναι ο βασικός μου στόχος. Να μην το παρατείνω αλλά να το τερματίσω το ταχύτερο δυνατόν. Τώρα για τις αποζημιώσεις προς τα θύματα. Κάνουμε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια στον τομέα αυτό για την επανόρθωση των ζημιών που υπέστησαν τα θύματα. Όπως είπαμε είναι 470.000 θυμάτων που έχουν τύχει επανόρθωση, αλλά ο συνολικός αριθμός είναι 6 εκατομμύρια. Ήταν τεράστιο το κόστος για τον προϋπολογισμό μας. Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ισταρία που δίνει επανορθώσεις στα θύματα προτού αποζημιώσεις, προτού τελειώσει η σύγκρουση, η στρατιωτική. Πρέπει να έχει και συμβολικό χαρακτήρα εξανάγκησε αυτή η επανόρθωση. Πόσο κοστίζει ένα παιδί, μια κόρη, κύριε Χάουιτ. Πόσο κοστίζει ένας πατέρας, μια μητέρα. Είναι αδύνατον να αποζημιώσει κανείς κάποιον για την απώλεια ενός οικείου. Γι' αυτό αυτές οι επανορθώσεις έχουν συμβολικό χαρακτήρα. Είμαστε σε μια οδομάτισης και έγινε μια μελέτη στο Χάρβαρτ που αφορά τη διαδικασία ειρήνευσης στην Κολομβία και αναφέρεται ότι είναι μια πρωτοφανής διαδικασία στην ιστορία αυτή. Σε συγκρούσεις όπως είναι η δική μας, μιλάμε για επανορθώσεις που στρέφονται προς το 14% του πληθυσμού, όχι το 1 ή 2% όπως σε άλλες περιπτώσεις. Εξακολουθούμε την προσπάθεια αυτή. Το ότι τα θύματα συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Μου λέτε, πώς μπορώ να φέρω 6 εκατομμύρια θυμάτων στην Αβάνα. Θα ήταν θαυμάσιο, αλλά φυσικά είναι αδύνατο να γίνει κάτι τέτοιο. Τι αποφασίσαμε λοιπόν για αυτό το λόγο. Κάποιοι αμερόληπτοι φορείς που να έχουν την εμπιστοσύνη και των δύο πλευρών. Η Εκκλησία, ο ακαδημαϊκός χώρος, τα Ηνωμένα Έθνη να μπορέσουν να επιλέξουν εκπροσώπους των θυμάτων για να μπορέσουν να εκφράσουν την άποψη των θυμάτων. Δεν μπορούμε όλα τα θύματα να τα φέρουμε. Αλλά νομίζω ότι υπήρξαν εκπρόσωποι από όλη την κοινότητα των θυμάτων που επελέγησαν με αυτόν τον τρόπο. Ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστέψτε με, κύριε Χάουιτ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Κολομβία έχει κάνει τεράστιες πρόοδους στον τομέα αυτό σε ό,τι αφορά την πολιτική μας για την, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Σύνταγμα μας είναι από τα συντάγματα που δίνουν τις περισσότερες εγγυήσεις <clears throat> σε παγκόσμιο επίπεδο. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες σε όλους τους τομείς που μας έχουν βγάλει από τη μαύρη λίστα σε πάρα πολλούς διεθνείς οργανισμούς. Δεν είναι ότι η χώρα μας είναι παράδεισος εξακολουθούν να υπάρχουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξακολουθούν να υπάρχουν δολοφονίες συνδικαλιστών αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάθε φορά μειώνονται, κάθε φορά μειώνονται και κανείς δεν μπορεί να πει πια ότι όλα αυτά είναι πολιτική, στρατιωτική, είναι πολιτική κρατική. Εξακολουθούν να υπάρχουν βέβαια ομάδες οι οποίες προβαίνουν σε αντεκτικήσεις, κάνουν αυτόνομες ενέργειες, αλλά αυτή τη στιγμή διώκονται με αμήλικτο τρόπο από το κράτος και τη δικαιοσύνη. Μπορείτε να πείτε ότι μια δολοφονία συνδικαλιστή είναι ήδη μια δολοφονία πέρα από ό,τι θα έπρεπε να συμβαίνει. Έχουμε προσπαθήσει να μειώσουμε το κόστος της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κόστος της προστασίας των συνδικαλιστών και των αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι. Μου λέτε γιατί το κάναμε αυτό. Έχουμε μειώσει πολύ περισσότερο τον προϋπολογισμό σε άλλους τομείς, σε τομείς που έχουν να κάνουν με την πολιτική, με την προστασία πολιτικών που ζητήσαν συγκεκριμένα προστασία από ό,τι των ε, αγωνιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συνδικαλιστών. Η προστασία αυτή είναι ένα έθιμο το οποίο είναι ιδιαίτερα πολυδάπανο. Έχουμε τόσους ένοπλους φρουρούς οι οποίοι παίζουν το ρόλο των σωματοφυλάκων. Σιγά σιγά προσπαθούμε να φέρουμε σε κάποιο λογικό επίπεδο αυτή την προστασία για όλους. Αλλά η προστασία αυτή δίδεται σε αυτούς οι οποίοι χρειάζονται μια τέτοια προστασία, πιστέψτε με. Ο κύριος Τάνοκ. Σας ευχαριστώ για τα ερωτήματά σας. Η πολιτική για τα ναρκωτικά. Πριν από δύο-τρία χρόνια, όταν ήμουνα ήδη πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρότεινα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ναρκωτικών με μια διαφορετική προσέγγιση, με μια πιο σύγχρονη προσέγγιση. Η Κολομβία υπήρξε η χώρα και ξέρω σαν Κολομβιανός περί πρόκειται ήταν η χώρα που πλήρωσε το μεγαλύτερο τίμημα σε όλο τον κόσμο στον αγώνα αυτόν εναντίον των ναρκωτικών που πριν από 40 χρόνια κήρυξαν τα Ηνωμένα Έθνη. Χάσαμε τους καλύτερους ηγέτες μας, τους καλύτερους δημοσιογράφους μας, τους καλύτερους αστυνομικούς μας, τους καλύτερους δικαστές μας σε αυτόν τον αγώνα κατά των εμπόρων ναρκωτικών. Μπορέσαμε να εξαρθρώσουμε το καρτέλ του Κάλι, το καρτέλ του Μεντεγίν, των εμπόρων ναρκωτικών που πολλοί θεωρούσαν ότι ήταν ανίκητα, καταφέραμε να μειώσουμε την έκταση που καλλιεργείται με κόκα. Αλλά φαίνεται ότι όταν κάνει κανείς άσκηση στο ποδήλατό του, κοιτάζει δεξιά, κοιτάζει αριστερά και είναι στο ίδιο σημείο εξακολουθεί κανείς να μπορεί να πάρει κοκαίνη στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο, στο Μαϊάμ και στην Ποκοτά. Είναι πολύ εύκολο. Ο πόλεμος λοιπόν αυτός κατά των ναρκωτικών που κηρύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη πριν από 40 χρόνια φυσικά δεν έχει κερδιθεί. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι πρέπει να δούμε πού δεν πηγαίνει καλά η πολιτική μας και πού μπορούμε να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Γι' αυτό στη διάσκεψη κορυφή των χωρών της, ε, του Δυτικού Ημισφαιρίου Έκανα μία πρόταση που δέχτηκαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς και αυτή τη στιγμή συζητάτε αυτό το θέμα το οποίο 2016 θα έρθει και στα Ηνωμένα Έθνη για να δούμε τι άλλες νέες και πρωτότυπες πρωτοβουλίες θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο γιατί καμία χώρα από μόνη της θα μπορέσει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Οποιαδήποτε δράση η οποία έχει μονομερή χαρακτήρα θα έχει σαν αποτέλεσμα την αποτυχία. Δεν είναι δυνατόν παραδείγματος χάρη στην Κολομβίνα να πω σε ένα γεωργό σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Κολομβίας ότι θα το στείλω στη φυλακή γιατί καλλιεργεί μαριχουάνα όταν στο Κολοράδο στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι νόμιμο το να καλλιεργεί κανείς μαριχουάνα. Αυτές είναι αντιφάσεις οι οποίες δεν μπορούν να σταθούν. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε ε, την αντιμετώπιση μας σε παγκόσμιο επίπεδο για το πρόβλημα αυτό. Δυστυχώς εξακολουθεί το πρόβλημα αυτό να είναι σημαντικό και να... Για τη Βενεζουέλα τώρα και για τις άλλες γειτονικές χώρες. Η Ευρώπη γνωρίζει ότι ποια είναι η real πολλοί από τους γείτονές μας σκέφτονται με διαφορετικό τρόπο. Έχουμε διαφορετικούς στόχους, έχουμε διαφορετικά αναπτυξιακά πρότυπα, αλλά εγώ πιστεύω στις καλές σχέσεις γειτονίας με όλες τις χώρες του κόσμου, σεβόμενοι τις διαφορές μας και επιλύοντας τις διαφορές με διπλωματικό λόγο και όχι μέσω ύβρεων στα πλαίσια των μέσων ενημέρωσης λες και έχουμε να κάνουμε με εγώ θα ήμουν ε, δημόσιος ε, γνωστός εχθρός του Προέδρου Τσάβες. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να, ε, να οξύνουμε τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν και ότι προσπαθήσαμε με τον προηγούμενο πρόεδρο να έχουμε εγκάρδιες σχέσεις Νομίζω ότι προς όφελο και της Κολομβίας και της Βενεζουέλας και του συνόλου της περιοχής. Πρέπει να αναγνωρίσω ότι ο Τσάβες ήταν πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του στην αρχή αυτή της ερηνευτικής συμφωνίας και πρέπει να το αναγνωρίσω και να το παραδεχτώ. Ε, Για τον κύριο Βαντάλεν. πώς εμείς προσπαθήσαμε να μορφοποιήσουμε γενικά. Υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες την χάνουν πολιτικής αναγνώρισης θα έλεγα, η ΦΑΡΚ. Και υπάρχουν και κάποια υπόλοιπα των παραστρατιωτικών που αντιμετωπίζουμε σήμερα σαν εγκληματικές ομάδες. Δεν μπορούμε να έχουμε με αυτούς διάλογο πολιτικό. Αυτές τις ομάδες τις καταπολεμούμε, προσπαθούμε να τις αποσαφρώσουμε και να είσαστε βέβαιοι ότι θα νικήσουμε. Υπάρχουν οι υπόλοιπα λοιπόν από τη διαδικασία αυτή. Αλλά παρόλα αυτά εμείς στρέφουμε όλη μας την προσοχή και όλη μας την ενέργεια στην καταπολέμηση αυτών των εγκληματικών ομάδων που τροφοδοτούνται από, την, από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και είναι εκτός ΦΑΡΚ και εκτός του ΕΛΕΛΕΝΕ. Αυτές οι ομάδες έχουν ανεπαρκή στρατιωτικό έλεγχο στις περιοχές αυτές και δεν είναι σε θέση να διαπραγματευτούν εξ ονόματος των μελών τους. Απόδειξη είναι ότι όταν οι ΦΑΡΚ δήλωσαν μια μονομερή κατάπαυση του πυρός, το σεβάστηκαν αυτό και το σεβάστηκαν και όλα τα περιφερειακά μέτωπα. Κάτι το οποίο δείχνει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο ελέγχουν. Επόμενη ερώτηση για την κατασκοπία. Εγώ θα σας απαντήσω με μια ερώτηση. Πώς ελέγχετε στην Ευρώπη εσείς ε, τους hackers, αν γνωρίζετε μία λύση να μου την πείτε. Σήμερα το πρωί είδα στο Financial Times ένα άρθρο που έλεγε ο διευθυντής της αντικατασκοπίας στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι είναι ε, εντελώς ανεξέλεγκτοι οι hackers ουσιαστικά στην Ευρώπη. Λοιπόν, αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και εμείς ε, στην Κολομβία. Εγώ ίδιος ήμουν θύμα. Παραβίασαν τον προσωπικό μου υπολογιστή και δημοσίευσαν τα προσωπικά μου ε, ηλεκτρονικά ταχυδρομεία. Δεν είχα δευτυχώς κάτι το μεμπτό. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Καλή ερώτησή σας, λύση εγώ δεν έχω στην παρούσα φάση. Λοιπόν αυτά. Α, μια μια στιγμή. Ούρτασουν. για την Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Ίσως να έχουμε κάποιες διαφορές ε, ε, διαρθρωτικού τύπου αν θέλετε. Εγώ πιστεύω στις ελεύθερες συναλλαγές και στο ελεύθερο εμπόριο. Πιστεύω ότι το ελεύθερο εμπόριο είναι παράγων ανάπτυξης. Μιλήσατε για τους παραγωγούς του καφέ. Ε, όχι λόγω της συμφωνίας αυτής, αλλά νομίζω ότι η παραγωγή του καφέ στην παρούσα φάση περνά την καλύτερη φάση στην ιστορία τους εξάγουν όλες τις ποσότητες του καφέ που επιθυμούν στην Ευρώπη, η οποία ευτυχώς τον καταναλώνει. Και ξέρετε ότι υπήρξε μια περίοδος ξηρασία στη Βραζιλία, κάτι το οποίο οδήγησε στην αύξηση των τιμών και έγιναν επενδύσεις στην Κολομβία για την μεγαλύτερη παραγωγή, για αύξηση της παραγωγής. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό ε, να διατηρήσουμε την ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές, να είναι ανοιχτή η πρόσβασή μας στις αγορές. Οι ελεύθερες συναλλαγές είναι κάτι το θετικό. Οι χώρες οι οποίες εντάσσονται σε διαδικασίες ελευθέρου εμπορίου αναπτύσσονται πολύ πιο γρήγορα από τις χώρες οι οποίες λειτουργούν με προστατευτικό τρόπο. Αυτό έχει φανεί στην Νότια Αμερική, στις χώρες της Νότιας Αμερικής. Η Συμφωνία του Ειρηνικού, οι χώρες που μετέχουν είναι φίλες του ελευθέρου εμπορίου, μειώνουν τα εμπόδια τα εμπορικά και γι' αυτό έχουν ρυθμούς ανάπτυξης οικονομικούς πολύ μεγαλύτερους από τις χώρες οι οποίες ε, κλείνουν τις οικονομίες τους. Είναι μια βασική προϋπόθεση για την ευημερία της κοινωνίας, μεγαλύτερη ανάπτυξη και δίδει φυσικά και περισσότερους πόρους για επενδύσεις στον κοινωνικό τομέα. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μπόρεσα να ανταποκριθώ στις ε, ενδιαφέρουσες ερωτήσεις τις οποίες μου απίφθηναν ε, τα μέλη της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για τους συναδέλφους που δεν μπορέσαν να λάβουν το λόγο. Πολλοί Ισπανοί φίλοι δεν μπορέσαν να λάβουν το λόγο. Παρ' όλα αυτά έχουμε ξεπεράσει κατά μισή ώρα τον προβλεπόμενο χώρο και έχουμε και το γεγονός ότι ο πρόεδρος δεν μπορεί να είναι αιώνια μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ελπίζω θα υπάρξει η ευκαιρία να συνεχίσουμε και στο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω και την Υπουργό Εξωτερικών η οποία ήρθε και αυτή να συμμετέχει στη συζήτηση αυτή. Παρακαλώ καθίστε μια στιγμή. Καθίστε παρακαλώ. Ελπίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε με την ε, κυρία Υπουργό Εξωτερικών τη συζήτηση στο μέλλον και να εμβαθύνουμε περαιτέρω για όλα αυτά που συζητήσαμε με σας κύριε Πρόεδρε και ελπίζω ότι η διαδικασία ειρήνευσης θα προχωρήσει με αίσιο τρόπο και γι' αυτό έχετε την απόλυτη υποστήριξή μας. Κάθε καλή τύχη σας ευχόμαστε γι' αυτό.